κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, το αρχικό κείμενο, τμήμα 1, ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αυτό θέλει έλεγχο, αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι, λίγοι, εγκρίθηκε. Παράγραφος 15 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Σε έξι τμήματα ονομαστικά το καθένα αρχίζει τώρα για το πρώτο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο πάντα ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται το τρίτο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφ... Πέρας. Εγκρίνεται. Το τέταρτο τμήμα, αρχής ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το πέμπτο τμήμα, αρχής ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το έκτο, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 17 σε δύο τμήματα. Πρώτον υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Σε 7 τμήματα όλα ονομαστικά. Πρώτη ψηφοφορία αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το τέταρτο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το έκτο. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και το έβδομο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 ονομαστικά αρχίζει τώρα. Ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το αρχικό τμήμα κείμενο καταπίπτει 21. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, ονομαστικά πάντα, αρχίζει τώρα, τμήμα πρώτο, παράγραφος 21. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 22 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Παράγραφος 23 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 24. Σε τέσσερα τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Υπέρ λέω. Το, κατά. Αυτό θα το ελέγξουμε λοιπόν. Αρχίζει ο έλεγχος για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 24. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα της ίδιας παραγράφου υπέρ κατά άποχες. Μάλλον έχει εγκριθεί, αλλά χρειάζεται παρόλα αυτά έλεγχο. Ελέγχουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Το τρίτο τμήμα ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το τέταρτο τμήμα ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 25, το αρχικό κείμενο, είπε κατά, άποχες, εγκρίνεται. Παράγραφος 26, το αρχικό κείμενο, είπε κατά, άποχες, εγκρίνεται. Παράγραφος 27 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο είπε κατά, άποχες, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές ε, απορρίπτεται. Τσεκ φωνές. Ωραία. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της 27. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 28 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 30 υπέρ κατά αποχές έλεγχος αρχής ψηφοφορία για την παράγραφο 30. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34 σε 3 τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η πέντε τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 11 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε το αρχικό κείμενο της 35, το οποίο όμως έχει καταπέσει. 36 παράγραφος, δύο τμήματα, ονομαστικά, τμήμα πρώτο, είπε συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονικά επίσης, η ψηφοφορία τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 37, το αρχικό κείμενο υπέ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 12, ονομαστικά, τροπολογία, η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η, παράγραφ... η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει το αρχικό κείμενο και πάμε στην παράγραφο 49 σε 5 τμήματα ονομαστικά το καθένα αρχίζει για το πρώτο ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα είπε; ε, Αρχίζει η ψηφοφορία, συγγνώμη. Ψηφίσατε όλοι. Τώρα ψηφίσατε όλοι. Ja, ist geschlossen. Πέρασε. Das ist angenommen. Εγκρίθηκε υπάρχει σφοδρά επιθυμία να μιλάω, ε, πιο αργά. Προσπαθώ, αγαπητοί συνάδελφοι, να τα αποκριθώ. Τρίτο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Abgelehnt. Απορρίπτεται το τέταρτο τμήμα. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το πέμπτο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 7 σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι με ονομαστική. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο δεν ψηφίζεται. 8 ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο ονομαστικά αρχίζει ψηφοφορία τώρα. Στην τροπολογία 8. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο έχει καταπέσει παράγραφος 58 σε δύο τμήματα του πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία, επαλήθευση. Haben Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Η εννέα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο έχει καταπέσει. 61 σε τρία τμήματα. Η παράγραφος πρώτο τμήμα ηλεκτρονική άρχεται. Και για τα τρία είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Abgelehnt. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Άρχη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφό 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 10. Υπέρ κατά άποχες αυτό θέλει έλεγχο αρχίζει τώρα για την παράγραφο 10 ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται λοιπόν το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πάντα ονομαστικά άρχεται για το πρώτο ψηφίσατε όλοι πέρας Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 67, το αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα ονομαστικά αρχίζει για το πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και το τρίτο τμήμα, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 70 το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, ονομαστικά τμήμα πρώτο αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 74, το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, το τμήμα πρώτον υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 76, το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο ονομαστικά αρχίζει ψηφοφορία τώρα. Για ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη α. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη β. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη για το λατινικό υπέ το πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη και υπέ το πρώτο τμήμα τους κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη εν. έχουμε την τροπολογία 3 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Ελέγχουμε την τροπολογία παριθμών 3, αρχίζει τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Α, εγκρίθηκε. Το αρχικό κείμενο καταπίπτει, αιτιολογική σκέψη O, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τη λατινικό σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη S, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα του ψηφίσματος ονομαστικά αρχίζει ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Wir kommen dann zum Bericht και τώρα περνάμε στην έκθεση της κυρίας Εράνθ Γκαρσία, ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα διενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος. Κυρία Ριβαζή, για τον ε, κανονισμό. Διαδικαστικό. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ενημερώσω, κύριε Πρόεδρε, του συναδέλφου ότι υπήρξαν σοβαρέ δυσλειτουργίε ό,τι αφορά αυτή την έκθεση. Γνωρίζετε ότι η έκθεση αυτή αφορά ε, τα επίπεδα ραδιενέργειας από τρόφιμα σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Ε, είχαμε προσκαλέσει εμπειρογνώμες από την Ευρατόμου. Δεν ήρθαν, δεν θέλησαν να έρθουν. Ζητήσαμε να μας κατονομάσει εμπειρογνώμονες, η Κομισιόν μας είπε δεν γίνεται να δώσουμε ονόματα. Όμως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία διακυβεύονται και γι' αυτό διακόπτεται Δυστυχώ ε, Δυστυχώς δεν ήταν επί της διαδικασίας το ερώτημά σας. Ξεκινάμε λοιπόν να μπλόκα με τις τροπολογίες ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Τροπολογίες 1 έως 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται ονομαστικά οι 5. Θέλετε να μιλήσετε. Όχι. Λοιπόν, ονομαστικά η τροπολογία 5 άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δύο τμήματα ή 7. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τη 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή 16. Δύο τμήματα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 55 ονομαστικά άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 40 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται 57 D. Ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το νομοθετικό ψήφισμα ονομαστικά τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Ήταν πολύ σαφές. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Μισό λεπτό. Εγκρίνεται. Κύριε Φόξ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να προτείνω να ε, ακολουθήσει η έκθεση Ρέντα για να αναβάλουμε τις υπόλοιπες ε, για το Σεπτέμβριο. Με την αδειά σας να σας εξηγήσω γιατί. Είναι παράλογο να έχετε 25 λεφτά ψηφοφορίας την Τρίτη και 2 ώρες την Πέμπτη για εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας και ψηφίσματα εκ των οποίων κανένα εκ των οποίων κανένα δεν επήγει. Και πρόεδρε, οι υπηρεσίες θα έπρεπε να κανονίζουν καλύτερα τις ψηφοφορίες. Θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες στην Τρίτη και λιγότερες στην Πέμπτη. Προτείνω λοιπόν να δούμε την εκτισερέντα στη συνέχεια και να αναβάλουμε όλα τα υπόλοιπα, όλες τις υπόλοιπες για το Σεπτέμβριο. Κύριε συνάδελφε Φόξ, θέλω να πω ε, και να αποκρούσω απολύτως, μια και διαπαντό ότι ευθύνονται οι υπηρεσίες γι' αυτό. Πρώτον, η ε, διάσκεψη των Προέδρων, εσείς δηλαδή αποφασίζει τη διάταξη των εργασιών και βλέπετε και στον κατάλογο ψηφοφοριών ε, ποιες είναι οι ψηφοφορίες. Αλλά αυτό καθορίζεται ε, ουσιαστικά από τον αριθμό των ε, κατατμήματα ψηφοφοριών και των ε, ε, χωριστών. Και εμείς δεν έχουμε βοηθούς στις υπηρεσίες ε, για να ξέρουν τι θα ζητήσουν. Μπορείτε τη διοίκηση να την κατακρίνετε, αλλά μην κάνετε bashing και bullying χωρίς λόγο στη διοίκηση. Εντάξει, κύριε Φόξ, ερμηνεύω έτσι αυτό που ζητάτε. Πρώτον, να ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση Ρέντα και τις υπόλοιπες να τις ε, αναβάλουμε. Άρα μάλλον έχει νόημα να κάνουμε δύο ψηφοφορίες. Συμφωνείτε ποιος συμφωνεί να ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση Ρέντα. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η, ε, το, ε, έτοιμά σας. Τσεκ, φωνές. Να το ελέγξουμε κιόλας. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Υποθέτω ότι δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για το δεύτερο αίτημα και συνεχίζουμε λοιπόν. Έκθεση για τη δημιουργία Ένωσης Κεφαλαιογορών. Η τοπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τρία ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται πέντε ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται τοπολογία 8 ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 9 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 11 ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κύμα της 50 ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παρά... Συγγνώμη, τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα τώρα όπως έχει τροποποιηθεί ή δεν το τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστικά ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Δεκτό. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια. Έχουμε από την Επιτροπή 9, τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές, 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπ ήταν μεν σαφές, αλλά στο επαληθεύσουμε. Τη 10 άρχεται ονομαστικά η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τροπολογία 10. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται τροπολογία 11 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. απορρίπτεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές, άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτό. Το 34. Άρα καταπίπτει το αρχικό κείμενο της 2. Στη 12 πάμε υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 5 αρχικό κείμενο ονομαστικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. Οι σοσιαλδημοκράτες να δίνουν έτσι κάποια ένδειξη παρακαλώ για να ξέρουμε τι γίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω απορρίπτεται αλλά να το ελέγξουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι, άρχεται ηλεκτρονικά. Για την τροπολογία 15. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι καθόλου σαφές να ψηφίσουμε ονομαστικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10, αρχικό κείμενο, δύο τμήματα, ονομαστικά πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. 37 τροπολογία, ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 38 ως προστίκη. Όχι αντικατάσταση. Ψήφι περ. Είναι περίπου τα ίδια βλέπω υπέρ και κατά, γι' αυτό να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο τους 12 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19 αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Παράγραφος 20 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 39 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 21 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 22 παράγραφος. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά αποχές και αυτό θα το ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 16 για υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 το αρχικό κείμενο της παραγράφου ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε για την ε, τροπολογία 2, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 26 αρχικό κείμενο σε δύο τμήμα πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 26. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Η ψήφι υπέρ. Να το ελέγξουμε και αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 ότι ονομαστικά άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 27 αρχικό κείμενο ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29 το αρχικό. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος, συγγνώμη, τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό της παραγράφου 31 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45 ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. εγκρίνεται. 46 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η, 20, η τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Νομίζω εγκρίνθηκε, αλλά να ελέγξουμε την 20 άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογή 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 35, αρχικό κείμενο ονομαστικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Angenommen. Antrag 22 dafür. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 23. Ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt. Die Abstimmung geschlossen. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 36 ε, το αρχικό κείμενο υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται. δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 ε, αρχικό κείμενο υπέρ σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα κατά Τι έγινε, αφήσαμε την 25. 25 περίφθη. 38 λέω. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Είναι σε δύο τμήματα. Κατά. Την 25 δεν την ψηφίσαμε. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρο, εγώ φταίω, ε, δεν είδα την 25. Ψηφίζουμε την 25 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 38 τώρα, το αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 41 ονομαστικά αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 40, το αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα είναι όλα ονομαστικά. Τμήμα πρώτο αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασα. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο λοιπόν καταπίπτει. Πάμε στην παράγραφο 46 υπέρ του αρχικού κειμένου. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 33 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 υπέρ, τροπολογία, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Παράγραφος 50, το αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρία τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 30 υπέρ, κατά. Αυτό θέλει έλεγχο, άρχεται η ψηφοφορία. Για στην τροπολογία 30. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Αιτιολογική σκέψη C, το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη D, το αρχικό κείμενο. Α, ε, έλεγχος για το C, το αρχικό κείμενο, επαλήθευση ηλεκτρονική, αυτού που μόλις ψηφίσαμε. Αιτιολογική σκέψη C. Ψηφίσατε όλοι. Παράθυρο. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην αιτιολογική σκέψη D. Ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 είπε. Κατά. Δεν βλέπω. Μια μεγάλη πολιτική ομάδα πια σταμάτησε να εκπέμπει υπέρ κατά αποχές α τώρα εγκρίθηκε κύριε Γκερέρο Έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η αιτιολογική σκέψη έτσι στο αρχικό κείμενο με ηλεκτρονική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι <laughs> Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 31 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, ε, ε το αρχικό κείμενο, επε, πατά. Άποχες. Απορρίπτεται τσεκ φωνές. Αρχίζει λοιπόν ο έλεγχος. Αιτιολογική σκέψη ε. Ψήφισατε όλοι. Συγγνώμη, Γιώτα, όχι έψη. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η ταπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 42 με ονομαστική κλίση. Τροπολογία αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά και αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Wer Ποιος ζητεί το λόγο. Die Abstimmung ist, το λόγο. Eröffnet. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία και όταν θα έχετε ψηφίσει όλοι θα κηρύξω και το πέρας. Εγκρίνεται. nun Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016. Το λόγο ζήτησε ο κύριος Γκερέρο. Κύριε Γκερέρο, έχετε το λόγο. Αλλά δεν, μπορεί, δεν ανάβει το μικρόφωνο σας τώρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα, Πρόεδρε, να ζητήσω η ψηφοφορία για το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναβληθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Με στόχο να προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμφωνία ε, πιο συνενετική και πιο αντιπροσωπευτική για τις κοινέ προτεραιότητες και ισορροπημένες προτεραιότητες των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκερέρο. Υποθέτω και θεωρώ ότι αυτό το ζητάτε εξ ονόματος της ομάδας σας. 90, Absatz 1 erfüllt und ich lasse... Είναι το αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού. 190 ε, εδάφιο 2 πρέπει να μιλήσει ένας υπέρ και ένας κατά. Ποιος θέλει να μιλήσει υπέρ. Ο συνάδελφος Eichhout. Ήδη τον Ιανουάριο ε, αποτύχαμε να ε, ψηφίσουμε ε, για το πρόγραμμα εργασίας του 2015. Θέλουμε να αποφύγουμε να επαναληφθεί αυτό το για το 2016. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την αναβολή της ψηφοφορίας για το Σεπτέμβριο. Ε, αυτός ήταν υπέρ. Άλλος κατά από άλλη πολιτική ομάδα ή δυνατόν, η συνάδελφος Φόρτ. Έχοντας προεδρεύσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων επί του θέματος, είναι ντροπή, μεγάλη ντροπή, ότι αποχωρήσαμε τη Δευτέρα το βράδυ από εκείνο το διαπραγματευτικό τραπέζι, ενώ οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ συμφωνούσαν ε, σε ένα κοινό κείμενο και ξαφνικά μια ομάδα αρνείται να υπογράψει τη συμφωνία. Δεν ξέρω τι έχουμε να κερδίσουμε αν επανέλθουμε το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φόρτ. Ψηφίζουμε λοιπόν ποιο συμφωνεί με την πρόταση του κυρίου Γκερέρο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Αγαπητέ συνάδελφε, το, ε, ζητάτε επαλήθευση, άρχεται επαλήθευση. Ήθελα να σας πω αγαπητέ συνάδελφοι ότι σας ακούω και πιο σιγά να μιλάτε, δεν πειράζει. Ε, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε λοιπόν. Και περνάμε στο ψήφισμα που αφορά την κατάσταση στην Ιεμένη. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα έξι πολιτικών ομάδων με ναι, παράγραφος 3 σε δύο τμήματα, τμήμα 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 έχει προφορική τροπολογία εδώ. Ο συνάδελφος Κόουσο Περμούη υποθέτω ότι έχει τυπωθεί κιόλας. Παρακαλώ κύριε Κόουσο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, παρουσιάσω την εξή τροπολογία στη 2. α Εκφράζει την ανησυχία του απέναντι στο έντονο εμπόριο όπλο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες χώρες της περιοχής και ζητεί ε, σχετικά να ελέγξει το Συμβούλιο εάν έχει τηρηθεί ε, η διάταξη που αφορά το εμπόριο και τις εξαγωγές όπλου και κατά πόσο τα κράτη-μέλη τηρούν ε, την λόγο κοινή θέση. Διαφωνεί κανείς με αυτό? Das sind 40. sehr, Herr. Πάμε πολύ αγαπητέ συνάδελφοι κόου Έχουν εγερθεί 40 και πλέον συνάδελφοι. Ψηφίζουμε λοιπόν την αρχική τροπολογία 40 υπέρ κατά ε, δύο, συγγνώμη. Πρόκειται για την τροπολογία 2. Υπέρ για να σηκώνονται όμως. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 3. Δεν βλέπω. Να το ελέγξουμε ό,τι θέλετε. Αλλά αν ζητάει τσεκ η ομάδα που δεν δείχνει πώς ψηφίζει, δεν είναι πάρα πολύ αθλητικό το πνεύμα που σας διέπει. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 3. 3. Όχι 2. 3. 3. Γιατί γράφει 2 το μηχάνημα. Τη 2 την ψηφίσαμε. Es geht um den Änderungsantrag. Πρόκειται για την τροπολογία παριθμών 3. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η αιτιολογική σκέψη ε σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G υπέ κατά. Θέλει έλεγχο αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Είπε Στην αιτιολογική σκέψη H, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του, όπως τροποποιήθηκε, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην έκθεση παιδιών. Παράγραφος πρώτη σε εννέα τμήματα παρακαλώ. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το τέταρτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα είναι μονομαστική κλίση, τέσσερα επόμενα. Πέμπτο, άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το έκτο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το έβδομο, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται το 8, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Βέρας. Εγκρίνεται το 1, το τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Το αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά Υπέρ είστε ή κατά κύριε Φλέκενστάιν. Ξανά. Παράγραφος 13. Υπέρ. Κατά. Α, τώρα εγκρίθηκε. Παράγραφος 15. Σε τέσσερα τμήματα. Τσεκ. Ας το ελέγξουμε το 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15 σε τέσσερα τμήματα. Τμήμα πρώτο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά το δεύτερο αρχίζει τώρα η ψηφοφορία Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το τέταρτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19 το αρχικό κείμενο. Τσεκ θέλετε. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν το ελέγχουμε αμέσως. Στην τροπολογία 3 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Angenommen. Ε, εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέ. Κατά. Αποχέ Εγκρίνεται. Παράγραφο 25. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. Παράγραφο 44. Σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτον Ah, χαίρομαι που ο κύριο Γκερέρο δείχνει τι ψηφίζει και δεν δείχνετε εσεί. Λοιπόν, υπέρ, κατά. Στο 44-1 είμαστε. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η 49 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνονται. Η αιτιολογική σκέψη καίει υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά άρχεται τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάω στην έκθεση Κουκάν. Παράγραφος τέταρτη. Αρχικό κείμενο, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο, ονομαστικά αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκτη παράγραφος, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 με προφορική τροπολογία του κυρίου Κουκάν. Όχι, δεν έχει προφορική. Έχει. Ναι, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ μικρή τροπολογία στην 7η παράγραφο, η δεύτερη γραμμή, η λέξη for διαγράφεται και αντί γι' αυτό λέει redrilling. Ε, καλεί δηλαδή τον αντιπρόεδρο, την αντιπρόεδρο και είπατε εκπρόσωπο να προχωρήσει συνεργασία για την, με τους πραγματικούς Ευρωπαίους γείτονες με βάση τα πρότυπα κτλ. κτλ με τους, ε, ε που θέλουν willing και όχι really. Λοιπόν, ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ας το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία στο δεύτερο τμήμα της ενδεκάτης παραγράφου. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. Δεκατέσσερα δύο τμήματα. Πρώτο, ονομαστικά, αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο υπέρ. Ονομαστικά μάλλον. η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Είκοσι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 26 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα της 26. η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 31 ονομαστικά παρακαλώ, αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. πέρας Εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 δύο τμήματα το πρώτο παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 δύο τμήματα πρώτο παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο ονομαστικά να αρχίσει η ψηφοφορία Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται τροπολογία πρώτη ονομαστικά και πάντα ε, και σε δύο τμήματα. Αρχίζει το πρώτο τμήμα και η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 58 στο αρχικό κείμενο, σε τρία τμήματα το πρώτο ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικό L, λάμδα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Π, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά Αποχές απερίφθη το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Έκθεση Ρέντα. Παράγραφό 7 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα θα το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Αρχίζει προφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παρέφος 10, δύο τμήματα. Πρώτο παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 11 δύο τμήματα. Πρώτο παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Δεν είναι πολύ σαφές. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Το 13 σε 3 Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο υπέρ. Επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα. 13-2 αρχίζει η ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19 δύο τμήματα υπέρ, στο πρώτο, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21 σε δύο τμήματα. Το πρώτο κατά άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 27 της συναδέλφου Χάνιμπολ, πληροφορική τροπολογία. Κυρία Χάνιμπολ, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω στο τέλος της παραγράφου αυτή. Πιστεύει ότι οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί αποκλειστικά θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση όσον αφορά τις αμοιβέ βάσει διαπραγματεύσεων. Οι δημιουργοί πρέπει να μπορούν να αμείβονται για το περιεχόμενο που συνήθως είναι μουσική και περιορίζεται στο διαδίκτυο. Υπάρχουν αντιρρήσει στην κατάθεση προφορική τροπολογία. Das sind genug. Sie brauchen, können sitzen bleiben. Ε, εντάξει, καθίστε, καθίστε, φτάνει. Οπότε δεν χρειάζεται και ψηφοφορία. Και πάμε στην 28. Παράγραφος 28, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 38 αρχικό κείμενο, δύο τμήματα, το πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο ονομαστικά, αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται το 40 σε τρία κομμάτια, το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τρίτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 δύο τμήματα. Παρακαλώ. Ψηφίσαμε το 40 στο τρίτο τμήμα, το τρίτο τμήμα του 40 λέει ο πρόεδρος. Τρίτο τμήμα του 40. Μα, και να φωνάζετε δεν αλλάζει τίποτα. Να σας το εξηγήσω προσπαθώ. Forty five are three parts, and forty are indicated as three parts, and forty five are three parts. Nein, wir, ich habe hier einen dritten Teil. Ναι, υπάρχει ένα τρίτο κομμάτι που λέει, υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τις ε, σχετικές εξαιρέσεις. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι. Το ψηφίσαμε. Βλέπω ότι και το ΕΛΚ συμφωνεί και άλλοι. Για συνοηθείτε λίγο με τις υπηρεσίες σας. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 45 δύο τμήματα, πρώτο, υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραφώς 46, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές επερίφθη αρχικό κείμενο. Επαληθεύουμε την τροπολογία υπαριθμών 3 αρχίζει η ισοφορία. Έφυσαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 46 αρχικό κείμενο ονομαστικά. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 51 δύο τμήματα πρώτο. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 53 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 δύο τμήματα. Στο αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 59 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη, αιτιολογική σκέψη 1 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1, συγγνώμη. Επαληθεύω την τροπολογία 1. Τροπολογία 1 αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Κύριο Σάρβαμα, για το, επί του κανονισμού δηλαδή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο Πρόεδρος κάνει εξαιρετική δουλειά το απόγευμα. Προσπαθεί να κινηθούμε το ταχύτερο δυνατόν. Υποθετήστε ότι δεν θέλετε να περάσουμε όλη την πέμπτη το απόγευμα εδώ στη Μικύκλιο. Θα ήθελα να ρωτήσω από όλου να σηκώνουν τα χέρια τους όταν ζητά ψηφο ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα την 67 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ονομαστικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρα. Εγκρίνεται δεύτερο ονομαστικά. Αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα. Εγκρίνεται. Ε, σκέψη G, Z, υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Ο μικρόν σε δύο τμήματα το πρώτο παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη Ερ Ρο. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά αρχίζει ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. και εγκρίνεται. Έκθεση JIP. Εναλλακτικό καταρχάς έτοιμα πρόταση ψηφίσματο με την τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Αρχικό κείμενο τώρα, παράγραφο 25, σε δύο τμήματα. Ονομαστικά το πρώτο τμήμα αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 σε δύο τμήματα, πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 44, δύο τμήματα, το πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη τη λογική σκέψη Κ, τροπολογία πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε στο σύνολό του ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται προτελευταία έκθεση, ψήφισμα για την κατάσταση στον Μπουρουντή. Εφτά ομάδες έχουν συντάξει την πρόταση. Προφορική τροπολογία για την παράγραφο 2 έχει καταθέσει ο κύριος Μισελ. Έχει ανακοινώσει μάλλον. Κύριε Μισελ, αν έχετε το καλοσύνη από το μικρόφωνο. Ναι, έχω προφορική τροπολογία που πιστεύω ότι ενημερώνει το κείμενο γιατί οι εκλογές στο Μπουρούντι έγιναν. Προτείνω λοιπόν να αντικαταστήσουμε εκεί που λέει ότι ανησυχεί σοβαρά από το καταδικάζει. Υπάρχουν αντιρρήσει. Όχι. Ψηφίζουμε την παράγραφο 2 με τη μορφή αυτή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψήφισμα για τη Σεμπρένιρτσα. Κοινή πρόταση 5 ομάδων μετά την παράγραφο 6 προφορική τροπολογία του, κυρίου Γιάκοφτσιτς. Παρακαλώ. Θέλω να σας ζητήσω να στηρίξετε δύο προφορικές τροπολογίες, διότι χτες πάρθηκαν δύο αποφάσεις, δύο γεγονότα που πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στο ψήφισμά μας. 6α λέει, ελυπάτε που το Σεβούλιο Ασφαλείας που έχει την κύρια ευθύνη για την ε, ασφάλεια διεθνώ απέτυχε να περάσει ψήφισμα όσον αφορά τη γενοκτονία στη Σεβδένιτσα. Είναι ένα θλιβερό γεγονό μια που το Διεθνέ Δικαστήριο και ο ΙΕ έχουν πει ότι έγιναν τα εγκλήματα στην Σεβδένιτσα και πρόκειται για γενοκτονία. Αυτή είναι η πρώτη προφορική τροπολογία. Δεύτερη, καλωσορίζει την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας Εζεγοβίνης που λένε ότι 11 Ιουλίου είναι η μέρα Πένθους και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Υπερψηφίστε τα. Gibt es Einwände? Αντιρρήσεις υπάρχουν. Καλώς. Ψηφίζουμε λοιπόν με την προφορική τροπολογία. Παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ θερμά. Wir haben das jetzt in 84 Minuten geschafft. Τα καταφέραμε μέσα 48, 40, μέσα 84 λεπτά. Ε, θα μπορούσαμε ίσως να είχαμε κερδίσει και λίγο χρόνο περισσότερο αν σηκώναμε το χέρι πιο καλά. Λοιπόν, παρακαλώ